να ξεκινήσουμε αμέσως με την ημερήσια διάταξη. Το πρώτο σημείο αφορά την έγκριση αυτής. Όπως όλοι γνωρίζετε, η διαδικασία ορισμού των Ευρωπαίων Επιτρόπων και των χαρτοφυλακίων τους δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, οπότε η Επιτροπή δεν θα μπορέσει να προχωρήσει στην έγκριση των γραπτών ερωτηματολογίων και έτσι θα σας προτείνω να αναθέσετε στους συντονιστές δια γραπτή γραπτής διαδικασίας τη διαδικασία ε, των ερωτήσεων για τις ακροάσεις των επιτρόπων και αν δεν έχετε αντιρρήσεις μπορούμε να εγκρίνουμε την σημερινή μας ημερήσια διάταξη. Δεν έχετε παρατηρήσεις. Να περάσουμε τότε στις ανακοινώσεις των συντονιστών. Πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση όσον αφορά τον κανονισμό ε, για, τις, ε, για τα επιθετικά ε, ξένα είδη. Ε, αυτή η διόρθωση, ή μάλλον αυτός ο κανονισμός υιοθετήθηκε σύντομα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά η μαλλον αυτος ο κανονισμος υιοθετηθηκε συντομα απο το ευρωπαικο κοινοβουλιο αλλα η διασυνη και το κλείσιμο της θητείας, η ολοκλήρωση της θητείας δεν μας έδωσε αρκετό χρόνο στην ε, γλωσσική νομική υπηρεσία για να μπορέσει πριν από την τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια να περάσει στις απαραίτητες, να προβεί μάλλον στις απαραίτητες διορθώσεις. Γι' αυτό και οι διορθώσεις αυτές οι οποίες ε, έχουν γίνει θα πρέπει να εγκριθούν με την επόμενη Ολομέλεια. Εάν δεν υπάρξουν ε, παρατηρήσεις για αυτό το διορθωτικό μέχρι το τέλος της μέρας σήμερα, ε, τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Η δεύτερη ανακοίνωση αφορά την ε, διερμηνία σήμερα. Έχουμε 21 γλώσσες και ως ήθιστε αναμεταδίδεται η σημερινή συνεδρίαση στο web stream. Και μπορούμε να περάσουμε τώρα στο επόμενο μας σημείο που αφορά την ψηφοφορία. Καταρχήν, γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για τον προϋπολογισμό 2015 για όλα τα τμήματα. Εγώ είμαι ο εισηγητής, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω καμιά εισαγωγή. Να σας πω μόνο ότι θα ψηφίσουμε πρώτα το τμήμα που σχετίζεται με τους αριθμούς και στη συνέχεια, όπως είναι και το σωστό, θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση που έχουμε συντάξει. Θα ξεκινήσω λοιπόν αμέσως με την ψηφοφορία. Αν είστε έτοιμοι λοιπόν, θα ψηφίσουμε διανατάσεις της χειρός και αν είναι απαραίτητο θα κάνουμε και επαλήθευση ηλεκτρονική. Τώρα, ε, περνάμε λοιπόν στην τροπολογία του εισηγητή, 6.300, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερη. Εκχαούτ 63-34. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Όχι. Α, συγγνώμη. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Ideva anch'io. No, è Εγκρίνεται. Α, Πρώτα να πούμε ότι κλείνει η ψηφοφορία, ολοκληρώνεται. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Τροπολογία 163-33. Κάποιος διακόπτη. Πρόεδρε, εδώ το μηχάνημά μου και η κάρτα μου δεν λειτουργεί. Μπορείτε να στείλετε κάποιον τεχνικό. Eh, come vota lo contiamo, sì. non ci sono i tecnici come, come in plenaria. Possiamo solo chiedere al collega. Μπορούμε μόνο να σας ζητήσουμε να αλλάξετε θέση μαζί με την κάρτα σας να... για να δούμε αν έτσι λυθεί το πρόβλημα. Okay. Εμενταμέντο ΕΚΑΟΤ 6333. 6.333 εκχάουτ. Υπέρ, κατά. Αποχ... Εγκρίνεται. 63.32. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία του εισηγητή. 63.01 υπέρ κατά εγκρίνεται Τροπολογία Κονέτσινα Φερέιρα 6344 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία του εισηγητή 6302 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Τροπολογία του εισηγητή 6303 υπέρ κατά αποχές έγκρινεται. Τροπολογία Κονέσνα Φερέιρα 6338 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε, απορρίπτεται. Ναι, ναι, με συγχωρείτε, σαφώς απορρίπτεται. Κιόλας. Τροπολογία του εισηγητή 6305. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία Κονέστα Φερέιρα 6341. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία του εισηγητή 6304 περ. Κατά. απορρίπ, Ε, αποχές απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, με συγχωρείτε. 6306 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία του εισηγητή 6307 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία του εισηγητή 6308 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία ριβάζει 6336 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Κονέτσνα Φερέιρα 6344 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6345 Κονέτσνα Φερέιρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6346 Κονέτσνα Φερέιρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Νάντζι 6349 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Χολβένη 6350 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Καπούτο 6352 Υπέρα. κατά αποχές απορρίπτεται. Σας ζητώ να ψηφίσετε unblock από την 6309 μέχρι την 6313 του εισηγητή. Ε, υπέρ λοιπόν ποιοι είναι. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία ριβάζει 6337. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία Γκίγκολ Δεκχάουτε, 63-35, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63-14 μέχρι και 19 είναι ε, του εισηγητή και πρόκειται για αποκατάσταση του σχεδίου προϋπολογισμού. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 6347 Wilmot ε, και άλλοι. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6348 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία Γκάλολβένη 6351. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία Κάντενμπαχ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Εγκρίνεται. Τροπολογία του εισηγητή 6320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία Κονέτσνα Φερέιρα 6339 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία του εισηγητή 6321 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6322 του εισηγητή. Ποια είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63-40. Κονέτσνα Φερέιρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 63, ε, 23 και 24 μπορούμε να τις ψηφίσουμε από κοινού. Ποιοι ε, είναι υπέρ. Α, έχετε αντίρρηση. Εντάξει. Χωριστά λοιπόν. 63-23 πρώτα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63-24. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63-42 Κονέστα Φερέιρα ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα να δούμε αν μπορούμε να ψηφίσουμε ε, unblock από την 63-25 μέχρι την 6331. 31 την τελευταία. Ε, λοιπόν, 63-25 υπέρ. Κατά. Αποχές 6326 63-26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63-28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 63-29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63-31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε την γνωμοδότηση. Eh, Ξεκινάμε με την τροπολογία 1. Υπέρ ποιοι είναι. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές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 αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τώρα, τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti? Ε, ψηφίσατε όλοι. Το ΕΛΚ έχει δύο παραπανήσιους. Οπότε καλό δύο αναπληρωτές να μην ψηφίσουν. Πιπιέ, siete δύο di Από το ΕΛΚ είστε δύο παραπανήσιοι. Έχει... Okay. The vote is closed. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται... Συνεχίζουμε με ψηφοφορία. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένω, οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ακροάσεις των επιτρόπων προβλέπουν ότι κάθε υποψήφιος επίτροπος θα περιλαμβάνει τρεις γραπτές ερωτήσεις από πλευράς της Επιτροπής μας. Γνωρίζετε ότι η διαδικασία ε, ε, έχει καθυστερήσει και στην συνεδρίαση των συντονιστών αποφασίστηκε να προτείνουμε στην Επιτροπή να αναθέσει αυτήν την απόφαση στους συντονιστές για τα τρία γραπτά ερωτήματα που μπορούμε να διατυπώσουμε εκ των προτέρων. Θα πρέπει να επικυρώσουμε όμως αυτή την απόφαση με ψηφοφορία. Σας ρωτώ λοιπόν αν είστε υπέρ του να το αναλάβουν αυτό οι συντονιστές. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μάλιστα. Πλειοψηφία λοιπόν ε, το εγκρίνει. Και τώρα περνάμε στο σημείο το επόμενο. Στην εξέταση της ε, θέσης του Συμβουλίου θα δώσουμε αμέσως την, το λόγο στο Συμβούλιο για τη δυνατότητα ε, που μπορεί να έχουν τα κράτη-μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν ε, την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στις επικράτειές τους. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως στο Συμβούλιο, στην Ιταλική Προεδρία, ώστε να μας παρουσιάσει την θέση του Συμβουλίου. Στη συνέχεια βεβαίως θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Παρακαλώ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλους. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς Πρόεδρε και τα μέλη του Κοινοβουλίου για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε να σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο των κοινών θέσεων του Συμβουλίου για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η οδηγία για τη δυνατότητα περιορισμού ε, ή απαγόρευση της καλλιέργειας των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αποτελεί πραγματική νομοθετική προτεραιότητα για την Ιταλική Προεδρία και γι' αυτό το λόγο ελπίζουμε πως θα είναι δυνατόν να συνεργαστούμε μαζί σας με αποτελεσματικό τρόπο και στρέφαμε κυρίως ε, στην εισηγήτρια την κυρία και τους κοιόδης εισηγητές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία όσο γίνεται πιο σύντομα. Όπως γνωρίζετε, η συμφωνία ε, αυτή στο Συμβούλιο επετέχθη μετά από χρόνια τέλματος. Για χρόνια προσπαθήσαμε να βρούμε μια αποδεκ... ένα αποδεκτό συμβαστικό κείμενο ε, και μετά από πολλές προσπάθειες και αυτό το οφείλουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ελληνική προεδρία και ε, έτσι λοιπόν ε, καταφέραμε να βρούμε μια αποδεκτή, ένα αποδεκτό συμβαστικό κείμενο σχεδόν για όλα τα κράτη-μέλη, γιατί 27 κράτη-μέλη το υπερψήφισαν. Ο στόχος ο κύριος ε, αυτής της πράξης είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην απέτηση διατήρησης ε, του συστήματος ε, κοινοτικών αδειοδοτήσεων και ταυτόχρονα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει που έχουν πολλές χώρες αλλά και η κοινή γνώμη για μεγαλύτερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες οι εθνικές, οι περιφερειακές αλλά και οι τοπικές που σχετίζονται με τις διάφορες με διάφορα αίτια, βέβαια πολλά από αυτά σχετίζονται με την κοινή γεωρική πολιτική, αλλά χρειάστηκε λοιπόν, όπως σας είπα, μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί συμβιβαστικό κείμενο. Ε, στη βάση λοιπόν είναι η απέτηση ευελιξίας για τα κρατημέλη και μια αναφορά στην αρχή της επικουρικότητας που κατά τη γνώμη μας είναι αρχή που βρίσκεται στη βάση τις θέσεις του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση. Ελπίζουμε λοιπόν πως θα είναι μια, ε, ε, κάτι που θα σας βρει σύμφωνος, τουλάχιστον όσον αφορά τους βασικούς στόχους αυτού του κειμένου. Τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο περιεχόμενο της πρότασης, θα προσπαθήσω σύντομα να σας τους αναφέρω. Ε, το καινοτομία που εισάγει το Συμβούλιο είναι ένας μηχανισμός opt-out σε δύο φάσεις. Ο στόχος αυτού του μηχανισμού σε δύο φάσεις είναι να αναζητήσει την εγγύηση της μέγιστης νομικής βεβαιότητας από την αρχή. Δηλαδή σε μια πρώτη φάση το κράτος μέλος θα μπορέσει μέσω της Κομισιόν, δηλαδή με τη ε, διαμεσολάβηση της Κομισιόν, να ζητήσει από τον ετούντα μια έγκριση, δηλαδή βρισκόμαστε σε μια αρχική φάση της διαδικασίας αδειοδότησης, δηλαδή το κράτος μέλος μέσω της Κομισιόν θα μπορέσει να ζητήσει από τον ε, Τούντα να περιορίσει τη το γεωγραφικό εύρος της αδειοδότησης. Αυτό είναι μια πρώτη φάση που στόχο έχει να αναζητήσει κατά κάποιο τρόπο την εξέβρεση συμφωνίας εξ αρχής. Δηλαδή να εξαλείψει τα προβλήματα εξ αρχής, αν αυτό είναι δυνατόν. Και γι' αυτό και προβλέπεται ένα είδος ε, σιωπηρής ε, συνένεσης ε, που σημαίνει ότι το εύρος της διαδιοδότησης θα είναι εξ αρχής περιορισμένο. Δηλαδή θα περιορίζεται η γεωγραφική ε, κάλυψη. Αν δεν υπάρξει τέτοια συμφωνία, το κράτος μέλος θα έχει ωστόσο τη δυνατότητα παρόλα αυτά να περιορίσει και να απαγορέψει στην ε, επικράτειά του την καλλιέργεια των ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Και γι' αυτό το λόγο, και έτσι περνάμε και στο δεύτερο, στη δεύτερη φάση, όπου έχουμε ορισμένους όρους, κυρίως χρονισμού, έτσι ώστε να είμαστε ε, μάλλον να εγγυηθούμε την ε, ασφάλεια δικαίου, την ε, νομική βεβαιότητα για συγκεκριμένες επιτακτικές αποφάσεις. Όπως έκανε και το, Συμβούλιο, και το Κοινοβούλιο παλιότερα, το Συμβούλιο αποφάσισε να ακολουθήσει την ίδια δομή και να υποδείξει έναν μη εξαντλητικό κατάλογο, είναι ανοιχτό ο κατάλογος και αυτό είναι καλό να το υπογραμμίσουμε, ένα κατάλογο αιτίων με βάση τα οποία θα μπορέ... μάλλον, στα οποία θα μπορέσουν να αναφέρονται τα κράτη για να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν χορέψουν και όλα την καλλιέργεια. Θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε σε λεπτομέρειες την κοινή θέση, για παράδειγμα, ε, έχουμε βάλει πολλά, πολλά αίτια, ε, ας πούμε μιλάμε για στόχους κοινωνική, ε, γεωργικής πολιτικής, κοινωνικο-οικονομικά αίτια, το να αποφύγει η παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε άλλα προϊόντα. Έχουμε ένα μακρύ κατάλογο, αλλά είναι και ανοιχτός. Όσον αφορά άλλα στοιχεία, του κειμένου τη συμφωνίας είναι σημαντικό να σημειώσουμε μια διάταξη που βρίσκεται στο τέλος, μάλλον που επετεύχθη στο τέλος των διαπραγματεύσεων, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διοδότησης, δηλαδή και μετά από τη διαδικασία διοδότησης, μπορεί το κράτος μέλος σε περίπτωση που αλλάξουν οι αντικειμενικά οι συνθήκες να προχωρήσουν στην απαγόρευση και στον περιορισμό Εφαρμόζονται λοιπόν μουτάτες μουτάντες οι διατάξεις που σας περιέγραψα προηγουμένως για το opt-out και άρα το κράτος μέλος θα μπορεί και ακόμα και μετά την αδειοδότηση να προβεί στον περιορισμό ή απαγόρευση της ε, καλλιέργειας. Εξάλλου προβλέπονται όλα αυτά σε συμφωνία με τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για τις μεταβατικές διατάξεις ώστε να διέπουν τις διατάξεις που ισχύουν στην έναρξη της ισχύως αυτής της οδηγίας που ελπίζουμε ότι θα είναι όσο γίνεται πιο σύντομα και όσον αφορά την νομική βάση το Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει την νομική βάση που προτάθηκε αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώντας ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι η βασική ε, ο βασικός στόχος αυτής της πράξης. Τέλος και μια τελευταία παρατήρηση για την νομική μορφή της πράξης αυτής. Το Συμβούλιο, όπως θα δείτε, αποφάσισε να τροποποιήσει την νομική μορφή της πράξης, γιατί η Κομισιόν αρχικά είχε προτείνει κανονισμό. Ωστόσο, μετά από μια προσεκτική αξιολόγηση, το Συμβούλιο, σε συμφωνία με την Κομισιόν, αποφάσισε να μετατρέψει τον κανονισμό σε μια οδηγία γιατί θεωρούμε όντως ότι η μορφή οδηγίας είναι πιο κατάλληλη για ένα μέσο από το οποίο μπορεί να δώσει στα κρατημέλη τη δυνατότητα να αποφασίζουν κάτι και όχι να είναι ε, μια πράξη η οποία να είναι άμεσα εφαρμοστέα από πλευράς των ε, φορέων των, του χώρου. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Όπως γνωρίζετε, εμείς θα διαβιβάσουμε την κοινή γνώμη ε, επισήμως στο Ευρωκοινοβούλιο την κοινή θέση, με συγχωρείτε, ε, στην επόμενη Ολομέλεια, δηλαδή τη Σύνοδο της 15ης Σεπτεμβρίου, πράγμα που θα σημάνει την έναρξη της δεύτερης ανάγνωσης. Όπω είπα ήδη για την τελική Προεδρία πρόκειται για μεγάλη προτεραιότητα, αλλά θεωρούμε ότι και η κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια έδωσε τέτοια μηνύματα πολύ ξεκάθαρα, ότι δηλαδή τα θέματα αυτά είναι προτεραιότητα. Είναι θέματα τα οποία είναι προσφυλή σε όλη την κοινωνία, από τους ε, γεωργούς μέχρι τους καταναλωτές, γι' αυτό και θεωρούμε πως είναι πολιτική, πολιτικό μας καθήκον να ενεργήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα και ελπίζουμε ότι μαζί σας ε, με την κυρία Ρίση και τους ισχυώδεις ηγητές αλλά και, τους, ε, και, και όλους εσάς να μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε συμφωνία πριν το τέλος του Ελπίζω να ήμουν σαφής και ευχαριστώ και πάλι τον Πρόεδρο και όλους σας για αυτή τη δυνατότητα που μας δώσατε να παρουσιάσουμε και να δώσουμε το περιεχόμενο της κοινή θέση και εύχομαι καλή δουλειά σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Βεντουρέλη που στο όνομα του Συμβουλίου και της Ιταλικής Προεδρίας μας ενημέρωσε για αυτή την κοινή θέση του ε, Συμβουλίου. Τώρα πρέπει να διοργανώσουμε τις εργασίες μας, ε, να κάνουμε δηλαδή δύο γύρους ε, παρεμβάσεων. Ο πρώτος γύρος με τον εισηγητή καταρχήν και έπειτα την εισηγήτρια με συγχωρείτε και έπειτα με τους κοιόδης εισηγητές όπου θα έχουμε αρκετά ε, τίματα για χρόνο Στο τέλος του πρώτου γύρου ερωτήσεων θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου για να απαντήσει. Ε, δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στη συνάδελφο Φρεντερίκ Ρίς που είναι η εισηγήτρια για το Κοινοβούλιο ώστε να κάνετε δική της εισήγηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και δύο ερωτήσεις όμως, ε, παρακαλώ. Δεν έχουμε έγγραφο, πάντως... Μπορώ να κάνω τις δύο ερωτήσεις. Μπορείτε να μιλήσετε, να μας δώσετε τη θέση σας με την ησυχία σας και μετά ενδεχομένως αν έχετε και ερωτήσεις να κάνετε προς την Ιταλική Προεδρία μπορείτε βεβαίως να τις ε, υποβάλλετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Γιατί ναι, πράγματι ανέλησα κάπως την διαδικασία και σήμερα ναι μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα από το να θέσω ερωτήσεις. Έτσι κι αλλιώς ε, περιμέναμε πολύ καιρό για να φτάσουμε εδώ γιατί είχε μπλοκαριστεί η πρόταση αυτή στο Συμβούλιο για καιρό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε. Είναι πολύ σημαντική και οι διευκρινήσεις ε, της Ιταλικής Προεδρίας και είναι καλό που μπορούμε να ρωτήσουμε και το Συμβούλιο και την Επιτροπή για αυτή την πρόταση. Γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε να πούμε ότι στην Ευρώπη διαφέρουν οι απόψεις μας για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πολλές ε, προκαταλήψεις, αλλά υπάρχουν και απαιτήσει και η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου έδειξε πόσο αποκλίνουσες είναι οι απόψεις μας. Το σύστημα πάντως ξέρουμε ότι είναι τέτοιο που έπρεπε οπωσδήποτε να δοθεί μια διέξοδος, να πάψει πια αυτή η δυσλειτουργία όσον αφορά την ευρωπαϊκή αδειοδότηση που οδηγεί σε αδιέξοδα τις χώρες μέλη. Το ίδιο ισχύει και για τις απαγορεύσεις. Η Ιταλία το ξέρει και η Πολωνία. Η... Τα εθνικά δικαστήρια, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια καταδίκασαν πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι καλό, ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να αναλάβω μετά την Κορίν Λαπάς την έκθεση αυτή και να είμαι συγγήτρια. Είναι πολύ καλό να συνεργαστούμε καλά μεταξύ μας. Είναι ζωτική σημασίας για να προχωρήσουμε και να προχωρήσουμε για τα περισσότερα σημεία, το υπενθυμίζω αυτό, να έχουμε απόλυτες πλειοψηφίες. Είναι πολύ σημαντικό δεν είναι τυχαίο. Σε δεύτερη ανάγνωση, αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε το δικό μας στίγμα, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε ισχυρή πλειοψηφία για να περάσουν ε, τα σημεία εκείνα πάνω στα οποία συμφωνούμε. Τα βασικά σημεία ποια είναι. Εκείνα για τα οποία διαφοροποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η αιτιολόγηση. Αναφέρθηκε και η κυρία Ταρόλη. Γιατί, γιατί ο κατάλογος αυτός αιτιολόγησης είναι πολύ ε, πιο, φαίνεται πιο ωραία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν έχει δώσει μια πιο συγκεκριμένη λίστα, ένα κατάλογο με κατηγορίες, με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, με τις κοινωνικές και οικονομικές ε, περιπτώσεις, έχει να κάνει με τη χρήση γης, με την διευθέτηση του αγροτικού χώρου, τη χωροταξία κτλ. Βασιζόμαστε επίσης και σε επιστημονικά δεδομένα. Δεν είναι μόνο συμβολικό το θέμα, είναι πολύ ουσιαστικό και γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα τα κράτη-μέλη δεν θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα να έχουν τις δικές τους αντιρρήσεις και στα επιστημονικά συμπεράσματα. Υπάρχει η βάση 192 που δεν βλέπω το Συμβούλιο στη συμφωνία του να, το συμπεριλαμβάνει. Η πρόσωπος Ιταλικής Προεδρίας είπε ότι τώρα θα έχουμε κανονισμό και όχι οδηγία. Μα γιατί. Εντάξει, για να υπάρχει κάποιος παραλληλισμός, ε, ναι. Αλλά στην πραγματικότητα γιατί θέλουν κανονισμό αντί για οδηγία, τι υπάρχει από πίσω. Είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Γιατί δεν περιλαμβάνεται την νομική βάση 192 η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και επιτρέπει στα κράτη-μέλη να δίνουν περισσότερα επιχειρήματα για τους λόγους που τα οδηγούν να προβούν σε κάποια απαγόρευση. Ο κατάλογος των κριτηρίων, περιβαλλοντικών ε, κριτηρίων, είναι λοιπόν πολύ πιο συγκεκριμένο όπως έλεγα και πριν και με πολύ περισσότερα επιχειρήματα η δικιά μας. Και θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από το Συμβούλιο και την Επιτροπή τι εννοούμε με τον στόχο αυτό της ε, ΕΦΣΑ. Και έχουμε παραδείγματα. Σίγουρα θα υπάρξουν διάφορα σχόλια. Ο κρογωνιαίος λίθος είναι το πρώτο στάδιο, που είναι ένα νέο στάδιο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολα να το συγκρίνουμε με τα βιοκτόνα, Πρόκειται για μια καινοτομία και το καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν έχουμε ακολουθήσει αυτό το δρόμο άλλη φορά. Δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και γι' αυτό και υπάρχουν και πολλοί φόβοι που εκφράζονται για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί αυτό το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις χώρες που θέλουν να απαγορεύσουν και τις ευρωπαϊκές αρχές. Η Γαλλία ξέρω ότι δεν θέλει να βρεθεί απευθείας σε διαπραγμάτευση με τους κοινοποιούντες. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα παίξει τον ρόλο της του διευκολυντή, facilitator, στις διαπραγματεύσεις στο πρώτο αυτό στάδιο. Είναι μια διαδικασία που δεν την γνωρίζω καλά και μου βάζει πολλά ερωτήματα. Ανάλογα βέβαια με τις απαντήσεις, φαντάζομαι ότι θα μου δημιουργηθούν και άλλα ερωτήματα αργότερα. Έπειτα το θέμα του κατά πόσο είναι συμβατή η διαδικασία αυτή με τα κείμενα. Έρχομαι στην ουσία θέλουμε τα κράτη-μέλη, εφόσον το επιθυμούν, να μπορούν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Το θέμα των όρων, των προϋποθέσεων, γιατί η διαδικασία αυτή, το δεύτερο στάδιο, πρέπει να περάσει από τι διαπραγματεύσει. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε στο δεύτερο στάδιο αν προηγουμένω δεν έχουμε περάσει από το πρώτο που είναι οι διαπραγματεύσει. Γιατί όμω, Μήπω έτσι σε αυτό το δεύτερο στάδιο και αυτό είναι ο φόβο μου, αυτό το δεύτερο στάδιο που ήταν ο ο λίθος, γιατί περιλαμβάνει όλα τα επιστημονικά δεδομένα και λοιπά, όλα αυτά πάνω στα οποία δουλέψαμε πριν από τρία χρόνια, μπαίνει στο περιθώριο έτσι. Το πρώτο στάδιο γίνεται πιο σημαντικό. Αυτό είναι ο κίνδυνο για μένα. Υπάρχουν και δύο άρθρα τα οποία θα ήθελα να μου εξηγήσουν περισσότερο. Όλα είναι ουσιαστικά. Δεν είναι ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, όχι όλα είναι σημαντικά εδώ. Η συνύπαρξη των καλλιεργών είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα βιολογικά επίσης προϊόντα, όχι μόνο για τα παροδοσιακά. Και η οικονομική ευθύνη σε ποιον πάει. Η Επιτροπή τι λέει. Λέει ότι έχουμε ένα άλλο κείμενο του 2004 που αναφέρεται στην οικονομική ευθύνη. Ναι, ξέρουμε. Όταν όμως υπάρχει ζημιά σε βιολογικές καλλιέργειες, δεν αποζημιώνονται επαρκώς για τη ζημιά. Δεν έχει συμπεριληφθεί όμως κάτι εδώ για αυτό το θέμα. Είπα ότι θα κάνω δύο ερωτήσεις, ξέρω ότι έκανα πολύ περισσότερες, αλλά βασίζομαι και στους συναδέρφους για να κάνουν τις υπόλοιπες. Περιμένω τις απαντήσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ε, εισηγήτρια για αυτή την εισαγωγή στην ε, συζήτηση. Θα δώσω αμέσως το λόγο για το γύρο των σκιωδών εισηγητών και θα ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ και τη συνάδελφο Κόστιγκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και την Ιταλική Προεδρία για την παρουσίαση του συμβιβασμού επί του οποίου κατέληξε το Συμβούλιο. Ήδη η συγκήτρια κυρία Ρης τόνισε ότι από το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει την κατεύθυνση, έχει δώσει την κατευθυντήρια γραμμή και αν δούμε και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας βλέπουμε ότι αυτό που εκφράζεται είναι μια έντονη επιθυμία στην Ευρώπη για ένα πραγματικά στεγανό σύστημα του δικαιώματος αυτοδιαθέσεως όσον αφορά τις τεχνικές καλλιέργειας μεταλλαγμένων οργανισμών. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά το Συμβούλιο, έχουμε από την άλλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βλέπουμε ότι αυτό το ζήτημα της καλλιέργειας των σπόρων και βέβαια της ε, τεχνικής αυτής είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, είναι πραγματικά καυτό. Η διάθεση στην Ευρώπη γίνεται όλο και πιο αρνητική και κυρίως απέναντι σε διεθνείς ομίλους που κυριαρχούν στην αγορά σπόρων στην Ευρώπη. Έχει έρθει λοιπόν πραγματικά ο καιρός να υπάρξει πρόταση από το Συμβούλιο των Υπουργών για το πώς θα προχωρήσουμε. Προσωπικά θεωρώ τον συμβασμό που επιτεύχθηκε ως την δεύτερη καλύτερη λύση. Και η συγγήτριά μας άλλωστε τόνισε ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσει κάποιος, κάπως πιο περιοριστικά. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για σημαντική βελτίωση, δηλαδή ο συμβασμός αποτελεί βελτίωση. Βεβαίως στην Ευρώπη έχουμε συνηθίσει να ασκούμε την πολιτική των μικρών βημάτων. Αυτή η πρόταση μιας διαδικασίας σε δύο στάδια είναι γενικά αποδεκτή. Ακούσαμε και ορισμένες φωνές και μετά από την συμβαστική πρόταση του Συμβουλίου που ισχυρίζονται ότι αυτή η αίτηση η έγκριση για τη διάθεση στην αγορά ανοίγει πόρτες. Εγώ θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδίω και το Συμβούλιο Υπουργών να ξεκαθαρίσουν απόλυτα την νομική κατάσταση. Το Κοινοβούλιο έχει καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα βασισμένα σε κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Στη χώρα μου την Αυστρία υπάρχει μεγάλο μέρος του καλλιεργούμενου εδάφους το οποίο χρησιμοποιείται για βιολογική γεωργία. Όσοι λοιπόν απορρίπτουν την καλλιέργεια μεταλλαγμένων οργανισμών, μεταλλαγμένων, ε, μεταλλαγμένων φυτών, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν. Ακούγονται πολλές φωνές μεταξύ της κοινής γνώμης που θεωρούν ότι δεν είναι εξασφαλισμένο αυτό μέσα από την πρόταση. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην δεύτερη ανάγνωση του εγγράφου, να δούμε και τις διάφορες απόψεις που θα εκφραστούν ακόμη. Σε αυτό το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ε, γενετικής τεχνολογίας πρέπει να τοποθετηθούμε καθαρά και να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν χώρες μέλη οι οποίες δεν θέλουν τα μεταλλαγμένα, τους μεταλλαγμένους οργανισμούς στα χωράφια τους. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε στέρεες και γερά θεμελιωμένες λύσεις. Ευχαριστώ την κυρία Κόστιγκερ και τώρα για τους σοσιαλιστές ο Αντιπρόεδρος Μπαρνιό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να πω και εγώ δύο λόγια μετά από το Συμβούλιο για να πω ότι μια που είμαι συγητής από πλευρά των σοσιαλιστών να ξέρετε ότι πιστεύουμε πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα έχει να κάνει με ολόκληρη την ευρωπαϊκή κοινωνία. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 12ης Ιουνίου αποτελεί βέβαια ένα σημαντικό βήμα. Η πρόταση αυτή, το γνωρίζουμε, προσφέρει περισσότερη νομική ασφάλεια επιτρέπει να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη να περιορίσουν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους, όπως πολύ σωστά υπεθύμησε και η Φρεντερίκα Ρή, η συγγήτριά μα, και θα μπορούν στο μέλλον να επικαλεστούν νέους λόγους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, την παρουσία γενετικών, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε άλλα προϊόντα. Συνεπώς, για μας, και αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων έχει να κάνει με ερωτήσεις προς το Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο μας λοιπόν θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένο. μετά την απόφαση της 12ης Ιουνίου. Το κείμενο πρέπει να βελτιωθεί. Να έχουμε μια πραγματική δεύτερη ανάγνωση, ώστε Δεδομένων των όσων έχουμε ήδη πει πριν από τον τριμερή διάλογο και πριν από την ομόφωνη αυτή απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εμείς το Κοινοβούλιο να επιμείνουμε στις αποφάσεις μας. Το ερώτημα που πρέπει όμως να θέσουμε στους αυτούς μας είναι το κείμενο του Συμβουλίου δίνει αρκετά στέρεα νομική βάση προκειμένου να απαγορευτεί πραγματικά η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στις χώρες που το επιθυμούν. Και τι ρόλο παίζει η βιοτεχνολογία στις αποφάσεις που παίρνουμε. Και πρέπει να πάμε πιο μακριά ίσως για να διασφαλίσουμε την ελευθερία των χωρών αυτών που θέλουν να απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικά τροπομένων οργανισμών. Εμείς, σοσιαλιστές και δημοκράτες, έχουμε εδώ διάφορα ερωτήματα και προτάσεις που ήδη από σήμερα το απόγευμα θα υποβάλουμε γιατί σήμερα το απόγευμα θα συναντηθούμε με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Για παράδειγμα, να μπει στο συμβιβασμό και να μπουν νέοι ναι, λόγοι που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους. Να μην αμφισβητούνται στη συνέχεια από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για Εθνικές Αποφάσεις ή από τον ε, ΠΟΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Νομίζω ότι πρέπει εδώ πέρα να υπάρξει και ένα σύστημα αποζημίωσης εφόσον ε, υπάρξει ζημιά από καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Να ενισχύσουμε επίσης και τους κανόνες αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, της ΕΦΣΑ δηλαδή, που λαμβάνει η χώρα πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Και ξέρουμε, το είχε πει και η Κορίν Λαπάζ, η συγκήτριά μας την προηγούμενη θητεία, θα είναι δύσκολο να καλύψουμε τις ελλείψεις και να διευθετήσουμε με διαιτησία τις διαφωνίες που μπορεί να προκληθούν με την ΕΦΣΑ. Δεν πρέπει λοιπόν να διστάσουμε στα πλαίσια της δεύτερης ανάγνωσης να συμπεριλάβουμε πιο συγκεκριμένες διατάξεις. Και έτσι θα επιτρέψουμε η νομική αυτή ασφάλεια να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό επιθυμούμε να γίνει στην δεύτερη ανάγνωση που θα έχουμε στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Στάσης έχει το λόγο. να μέρους των Πρασίνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και με τις ερωτήσεις που έκανε η συγγήτριά μας που Είναι πολύ σωστές ερωτήσεις πιστεύω. Ιδιαίτερα όσον αφορά την νομική ασφάλεια. Εγώ δεν βλέπω γιατί το Συμβούλιο προσπαθεί να επιβάλλει τις απόψεις του στο Κοινοβούλιο. Η νομική βάση του άρθρου 192 είναι πολύ βασική και δεν βλέπω γιατί έχουμε απομακρυνθεί από την νομική αυτή βάση είναι ζωτική σημασία για μας. Στην πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων θέλω λιγάκι να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε. Στις 15 Ιουλίου ακούσαμε τον κύριο Γιούγκερ, ο οποίος αναφέρθηκε και στην νομοθεσία αυτή για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και είπε ότι οι διάφοροι κανόνες και διαδικασίες αδειοδότησης γενικά τροποποιημένων οργανισμών πρέπει να αναθεωρηθούν. Και είπε σαφέστατα ότι δεν θέλουμε πια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοδοτεί τέτοιους οργανισμούς όταν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο Συμβούλιο ε, Υπουργών δεν υπάρχει πλειοψηφία. Εφόσον λοιπόν είναι αυτό το πλαίσιο, σήμερα στην ανταλλαγή απόψεων πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και όλοι στο Συμβούλιο δεν θα υπάρξει αρκετή πλειοψηφία προκειμένου να εγκριθούν ε, διάφοροι γενετικά τροπομένοι οργανισμοί. Αντίθετα, διάφοροι θα καταψηφίσουν. Οπότε, εδώ γίνεται μια προσπάθεια αν θέλουμε πανεθνικοποίηση για το θέμα αυτό, κάποια κράτη θα είναι πάντα Κατά. Αλλά θα ξέρουν πάντα ότι μπορούν έτσι κι αλλιώς στις χώρες τους να απαγορεύσουν την καλλιέργεια των γενετικά τροπομένων οργανισμών. Υπάρχουν διάφορες λύσεις. Αν θέλουμε την επανεθνικοποίηση, τότε θα πρέπει να φροντίσουμε να μην οδηγήσει τα θέματα του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της ε, βιοπικιλότητας, όλα αυτά να αποδυναμωθούν και τελικά να αποφασίζονται στο Συμβούλιο Υπουργών και μόνο. Δεύτερον, πρέπει να φροντίσουμε η επικράτεια του κράτους μέλους που δεν θέλει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς να κατοχυρώνεται και νομικά. Γιατί διατυπώνονται φόβοι ότι έτσι όπως είναι διατυπωμένη η πρόταση δεν υπάρχει επαρκής νομική ασφάλεια. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να ε, μπορούν να καταδικαστούν από κάποιο δικαστήριο για την επιλογή τους αυτή. Γι' αυτό λοιπόν και το είπε και η συγγήτρια και το είπαμε και στην πρώτη ανάγνωση ότι πάνω σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε πολύ. Τρίτον, πρέπει να φροντίσουμε ότι οι αποφάσεις του Δεκεμβρίου του 2008 των Υπουργών Περιβάλλοντος να μην αποδυναμωθούν. Δηλαδή, το περιβάλλον να μετράει πάρα πολύ σε κάθε απόφαση που θα λαμβάνεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εγκριθεί και εμεί οι πράσινοι, όπως καταλαβαίνετε, θα επιμείνουμε πάρα πολύ σε αυτό. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια τροπολογία είναι ζωτική σημασία για να προστατεύσουμε το περιβάλλον γιατί υπάρχει το θέμα των ντομοκτώνων, των φαρμάκων γενικά. Η, έπειτα, η πρόταση του Συμβουλίου για τον ρόλο που παίζουν επιχειρήσεις στις αποφάσεις για μας είναι κάτι απαράδεκτο. Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε άδεια από τους γίγαντες των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και να λαμβάνεται υπόψη δικιά τους η άποψη στις αποφάσεις που θα παίρνουν οι ευρωπαϊκές αρχές. Έπειτα τα πρώτα δύο χρόνια λέει η πρόταση ότι μόνο θα μπορεί να υπάρξει αυτή η απαγόρευση. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχιστεί αυτό, να μην είναι περιορισμένο χρονικά. Και το τελευταίο μου σημείο, το έκτο, είναι, είναι το θέμα της ε, επιμόλυνσης από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Εδώ πρέπει να έχει κάποιος την ευθύνη πολλές χώρες ε, δεν έχουν καμία ρύθμιση για τη συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων και μη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Εδώ επίσης λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση και εμείς οι πράσινοι διαφωνούμε με την πρόταση που κάνει το Συμβούλιο και επιμένουμε στον συμβασμό στον οποίο δύσκολα καταλήξαμε σε πρώτη ανάγνωση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ σας είπα τι ανέφερε στις 15 Ιουλίου, οπότε περιμένουμε εδώ να τηρήσει τις υποσχέσεις του και η θέση του στην πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλουμε όσο γίνεται περισσότερο να διατηρηθεί. Τέλος, ελπίζουμε και προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία με τους σκιώδες εισηγητές και βεβαίως και με την εισηγήτρια ΡΙΣ. Ξέρουμε ότι έχει ανοιχτό πνεύμα και με τέτοιο πνεύμα θα γυριστεί και την υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Εκ μέρου τη ΚΟΕ, το λόγο έχει η κυρία Μπόιλαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Θα ήθελα πρώτα να την παρακαλέσω ωστόσο να αναπτύξει λίγο περισσότερο τα περί risk assessment γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε και ποιες είναι οι μακρόχρονες επιπτώσεις στην υγεία και στη βιοπικιλότητα, όπως έχει ζητήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω και συγκεκριμένες προτάσεις να κάνω για την κοινή θέση του Συμβουλίου. Ναι, μεν χαίρομαι που κατέληξαν έστω και με καθυστέρηση τριετίας στο κείμενο αυτό. Το κείμενο όμως το βρίσκω ασθενές και έχει και πολλά νομικά παράθυρα. Εξακολουθούν λοιπόν να υπάρχουν οι σχετικές δυσκολίες ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων. Η δυνατότητα των κυρίαρχων κρατών μελών να αποφασίσουν εάν θα περιορίσουν ή θα απαγορεύσουν την χρήση των GMO σε μέρος ή σε όλη την επικράτειά τους πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Και επομένως πρέπει η πρόταση να είναι πραγματικά στεγανή. Όπως είπα, υπάρχει ο κίνδυνος να στραφούν νομικά κατά των αποφάσεων αυτών, αυτών οι διεθνείς όμιλοι που εμπορεύονται τα GMO. Δεν συμφωνώ για παράδειγμα ότι οι χώρες μέλη για να μπορέσουν να απαγορεύσουν τα GMO πρέπει να ζητήσουν πρώτα από τους ε, διεθνείς ομίλους να μην τα διαθέσουν στο εμπόριο στην επικράτειά τους. Πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης λοιπόν και όχι να επιβάλλουμε το βάρος της αποδείξεως στις χώρες μέλη και να τις αναγκάσουμε να διαπραγματευτούν με τις εταιρείες όπου προφανώς υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Συμφωνώ επίσης με τις ανησυχίες των πράσινων και θέλω να δω η νομική βάση να φύγει από το άρθρο 114 και να πάει στο άρθρο 192 της συνθήκης. Να ληφθούν υπόψη τα πράγματα αυτά και οι νόμιμοι λόγοι ή θεμητοί μάλλον λόγοι για την απαγόρευση. Το άλλο που μας ενδιαφέρει είναι η μόλυνση από, μεταλλαγμένα, από μεταλλαγμένους σπόρους ή φυτά. Ακόμα δηλαδή και αν επιτυχώς απαγορεύσει μια χώρα μέλος στην καλλιέργεια των GMO στην επικράτειά της, εάν αυτό γίνεται σε μια γειτονική χώρα δεν υπάρχει καμιά προστασία. Διότι μπορεί να γίνει μόλυνση των φυτών από μεταλλαγμένα φυτά. Πρέπει λοιπόν να, υπάρξει, να υπάρξουν ε, ζώνες προστασίας ανάμεσα στα εδάφη εκείνα όπου καλλιεργούνται τα GMO και σε εκείνα όπου απαγορεύεται η καλλιέργειά τους. Έτσι λοιπόν δέχομαι μεν ως ένα πρώτο βήμα την ε, συμβαστική κοινή θέση του Συμβουλίου. Ελπίζω όμως ότι θα μπορέσουμε να εργαστούμε έτσι ώστε να την διορθώσουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Θα ήθελα σε αυτή τη φάση. Επειδή υπάρχουν ακόμα 7 ε, που θέλουν να πάρουν το λόγο, για να κλείσω και τον κατάλογο, θα ακούσουμε και αυτές τις ερωτήσεις και μετά θα δώσω το λόγο στην ε, Κομισιόν και στο Συμβούλιο για να απαντήσουν. Οπότε τώρα το λόγο να δώσω στον συνάδελφο Πέτερλε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις που πήραμε μέχρι τώρα. Τώρα μετά από τόσα χρόνια είμαστε πράγματι σε καλύτερη θέση. Θέλω έλεγα όμως επίσης ότι πρόκειται για ένα ζωτική σημασία θέμα στην ε, Σλοβενία πριν από τις εκλογές αλλά και μετά τις εκλογές συζητήθηκε πάρα πολύ. Κατά τη διάρκεια ακόμα και των διακοπών δεν μ' άφησαν ήσυχο είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ το κοινό. Είναι ένα από τα πιο βασικά θέματα που βρίσκεται στο μυαλό των ε, πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ που είμαι και μελισσοκόμος το γνωρίζω το πρόβλημα και με απασχολεί. Διαπραγματευόμαστε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ότι κάνει το θέμα που συζητάμε σήμερα ακόμα πιο σημαντικό. Παρά τις προσπάθειες για διαφάνεια, εξακολουθεί να υπάρχει δυσκολία όσον αφορά τη νομική ασφάλεια, το είπε και η κυρία και άλλοι. Συμφωνώ με όλες τις παρατηρήσεις και τις αμφιβολίες που ακούστηκαν. Λαμβάνοντα υπόψη λοιπόν όσα ακούω από τους πολίτες, έχω την αίσθηση ότι οι καλλιεργητές γενικά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θέλουν, ξέρουν από πριν πού θέλουν να δυσδύσουν και σε ποιες περιοχές θέλουν να έχουν τις καλλιέργειές τους. Και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί αυτός που δεν θέλει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς είναι αυτός που πρέπει να βρει επιχειρήματα για να αντιταθεί. Δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να έχουμε σαφή θέση για το ρόλο που θα παίξουν οι επιστήμη. Αν κάποιος έχει προκαταλήψει και δεν θέλει, κανένα ή θέλει, κανένα επιχείρημα δεν πρόκειται να τον πείσει. Αυτό είναι αλήθεια. Στην πολιτική όλα τα επιχειρήματα, ακόμα και τα μη λογικά παίζουν ρόλο. Και εδώ θα θυμίσω αυτό που είπε και ο κύριος Στάες, ότι στη φύση καλλιεργούνται γεννητικά τροποποιημένοι οργανισμοί, όχι στην ε, αυλή μας ή μέσα στο σπίτι μας. Η επιστήμη λοιπόν δεν μπορεί να πει πολλά, δεν έχει να πει πολλά όσον αφορά τις επιπτώσεις επιμόλυνσης από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, όταν αυτή μετά από χρόνια θα αρχίσει να φέρνει επιπτώσεις. Δεν τις ξέρουμε ακόμα. Πρέπει να έχει κανείς το δικαίωμα να πει όχι και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκές λύσεις γι' αυτό. Οπότε ανησυχώ με την έννοια αυτή της επανεθνικοποίησης. Πρέπει να παραμείνει ευρωπαϊκό το ζήτημα και πρέπει να προστατεύουμε τους λαούς μας, να είναι καλά στην υγεία τους και αυτός ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω επίσης να ξέρω και το εξή. Ποιες είναι, ποια είναι τα θέματα σύμφωνα με την Ιταλική Προεδρία όπου είναι αφισβητήσιμα νομικά. Συνάδελφος Μπόρτζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ένα πράγμα είναι σαφές και από αυτό πρέπει να αρχίσουμε. Ότι δηλαδή οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θέλουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στις χώρες τους. Αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψουμε. Δεν θα ήταν σωστό. Ούτε πρέπει να προσπαθούμε να περιορίσουμε την κυριαρχία των χωρών μελών με τις αποφάσεις που παίρνουμε. Γιατί τότε οι πολίτες θα έχουν ακόμα λιγότερη εμπιστοσύνη σε μας. Κάποιες χώρες μέλη επιτρέπουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και κάποιες άλλες δεν το επιτρέπουν. Κάποιες χώρες είναι πολύ έντονες όσον αφορά τις αντιρρήσεις τους. Και πράγματι ε, η πρόταση αυτή, παρά τις αδυναμίες που έχουν ήδη φανεί, προσπαθεί να αποφύγει νέες αδυναμίες. Οι χώρες μέλη πιστεύω ότι πρέπει να έχουν περισσότερο περιθώριο ελιγμών για να αποφασίζουν αν θέλουν ή δεν θέλουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στην επικράτειά τους. Αυτό θέλουν οι πολίτες που εγώ εκπρόσωπω εδώ. Συνεπώς, αμφισβητούμε αυτή την πρόταση και πιστεύω ότι η νομική βάση πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και να μπορούν να ληφθούν περιοριστικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο, πολύ περισσότερο από ό,τι προβλέπετε τώρα. Αν εγκριθεί η ρύθμιση αυτή ως έχει, τότε οι παραγωγοί θα μπορούν να αντιτεθούν στις εθνικές απαγορεύσεις να τις προσβάλλουν. οποίο θα δημιουργήσει μια πολύ περίεργη κατάσταση. Τέλος είναι αυτή η πρόταση πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση μεν, αλλά για να πετύχει τους πραγματικούς στόχους, τότε κάποια σημεία πρέπει να αλλάξουν. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η συνάδελφος Όνερμεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι το σκέφτηκα πολύ αν θα πρέπει δηλαδή να ζητήσω το λόγο γιατί είναι ένα, για μένα δυσάρεστο θέμα. Εδώ και 15 χρόνια ασχολούμαι με την τεχνική και την τεχνολογία της γενετικής και πραγματικά ακόμη είμαι αναποφάσιστη σχετικά με το πώς θα ψηφίσω. υπάρχουν στοιχεία υπέρ της κοινή θέσεως του Συμβουλίου, αλλά από επιστημονική άποψη, εγώ είμαι επιστήμων αγρονόμος, βρίσκω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία κατά. Καλό βρίσκω ότι με τη νέα οδηγία επιτέλους δείχνουν πραγματικά τι επιθυμούν οι χώρες μέλη, διότι αυτό ήταν το πρόβλημά μας όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ότι οι χώρες μέλη δηλαδή δεν τολμούσαν να εκφράσουν άποψη δημόσια για τους μεταλλαγμένους οργανισμούς. Και απλώς απήχαν από του να λάβουν θέση. Καλό είναι λοιπόν τώρα που έρχεται αυτή η οδηγία. Οι χώρες μέλη λοιπόν θα πρέπει να δείξουν τι θέλουν, ναι ή όχι, την ε, γενετική τεχνολογία, διότι μέχρι τώρα τα φόρτωναν στο ευρωπαϊκό επίπεδο διότι φοβούνταν τους πολίτες τους τους ίδιους, ότι οι πολίτες θα στραφούν αντίον τους δηλαδή. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα είναι καλό να προχωρήσει η οδηγία. Διερωτώ με όμως εάν η διαδικασία εγκρίσεων εάν η κατάσταση αυτή μετά από την οδηγία 2001-18 αν δηλαδή θα είναι πραγματικά οι χώρες μέλη διατεθειμένες να αποφασίσουν για την αδειοδότηση ή απόρριψη της αδειοδότησης επιμέρους γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών. Μέχρι τώρα, όπως είπα, είχαν μπλοκάρει την ε, πορεία αυτή. Και εκεί όπου μέμφωμε τις χώρες μέλη είναι ότι μέχρι τώρα ποτέ δεν ενημέρωσαν πραγματικά τον κόσμο για το περί τίνος πρόκειται. Ουδής γνωρίζει πραγματικά. Ρωτήστε τον κόσμο, ρωτήστε. Κανείς δεν ξέρει τι είναι πραγματικά οι μεταλλαγμένοι γενετικά οργανισμοί. Είναι πια ζήτημα ιδεολογίας του καθενός. Και αυτό κάνει και το, αριστερο, και το μάλλον, πράσινο άκρο του φάσματος και το κόκκινο του πολιτικού φάσματος. Τέλος πάντων αυτή είναι η πολιτική. Είπα αρχικά ότι από αντικειμενική άποψη είναι λάθος να προχωρήσει αυτή η οδηγία και γι' αυτό εξακολουθώ να είμαι αναποφάσιστη όπως εξήγησα διότι η οδηγία απελευθέρωσης τότε, αυτή που ανέφερα προηγουμένως, ρυθμίζει λεπτομερώς τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να εξετάζονται οι γενετικά μεταλλαγμένοι οργανισμοί σχετικά με την αδειοδότησή τους. Τότε τίθεται πάλι όλα τα θέματα αυτά. Είναι ασφαλείς οι οργανισμοί αυτοί για την υγεία ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος. Εκεί όμως απαντώνται τα ερωτήματα αυτά, διότι επιτρέπεται η ελευθέρωσή τους μόνο εφόσον είναι αυλαβής. Τώρα πιστεύω σε σχέση με την κοινή θέση του Συμβουλίου βρίσκω αυτό τον ανοιχτό κατάλογο των λόγων απόρριψης πραγματικά αστείο. Από αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου μέχρι τώρα, άκουσα δηλαδή ότι να λένε ότι θα είναι δύσκολο να βρεθούν οι λόγοι. Όχι, αντιθέτως, Αντιθέτως είναι γελίος ο κατάλογος αυτός διότι μπορεί να επικαλεστεί καθένας οποιοδήποτε λόγο, οτιδήποτε, έτσι ώστε να απαγορεύσει περιφερειακά μέσα σε μια χώρα μέλος ή και σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας μέλους να απαγορεύσει δηλαδή την αδειοδότηση. Και μιλάμε και πάλι ότι σύμφωνα με το 2018 μιλούμε για ε, γάμα μειόμικρον των οποίων επιτρέπεται η χρήση. τελικώς καταλέγουμε σε ένα αυθαίρετο καθεστώς. Και με τη νέα οδηγία το ίδιο θα είναι. Καλύτερα να πούμε ότι δεν θέλουμε. Τουλάχιστον τότε θα είμαστε ειλικρινέστεροι. αυτό ο ψευδοκατάλογος με ενοχλεί, διότι πρόκειται πραγματικά για ψευδοκατάλογο. Τώρα έχω και μία ερώτηση ωστόσο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γεγονό ότι οι χώρε μέλη έχουν συμφωνήσει τώρα να μην περιβάλλουν την νέα με τον μαρδία του κανονισμού, αλλά να προτιμήσουν την οδηγία. Αυτό για μένα οδηγεί στην σκέψη ότι ε, τι άλλο θα βάλουν μέσα στην οδηγία οι χώρες μέλη. Μήπως με την επέκταση της οδηγίας αυτής σε ορισμένες χώρες μέλη τελικώς να καταλήξουμε το, σε ενδοκινοτικό εμπόριο σε παρεμπόδιση μάλλον του ενδοκινοτικού εμπορίου με γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς. Διότι κάτι τέτοιο βεβαίως θα είναι αντίθετο με την ενιαία αγορά και θα αντιβαίνει και στο γράμμα και πνεύμα της 2001-18. Εν τέλει, πρόκειται για περιορισμό και το βρίσκω κρίμα διότι περιορίζεται και η ελευθερία ημών των Ευρωπαίων για την οποία τόσο υπερηφανευόμεθα η επιχειρηματική ελευθερία των αγροτών όσων θέλουν να καλλιεργήσουν γάμα μειομικρών. Βέβαια, οφείλει κανείς να σεβαστεί και την πλειοψηφία. Εγώ ίδια όπως σας δήλωσα δεν γνωρίζω τα θα ψηφίσω ακόμη. Μάλλον δεν θα αντιταχθώ, αλλά δεν ξέρω και αν θα υπερψηφίζω. Πάντως η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ την κυρία Σόμερ. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος Γιαβόρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι νέοι αυτοί κανόνες έχουν ως στόχο την ενίσχυση της εθνικής κυριαρχίας. Οι χώρες μέλη θα έχουν έτσι τη δυνατότητα να επιτρέψουν ή αντίθετα να απαγορεύσουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Όπως κατά το παρελθόν, όταν κάποιες χώρες ήταν ε, κατά των οργανισμών αυτών, ήταν δύσκολο να απαγορευτούν. Είναι κάτι ενδιαφέρον η πρόταση αυτή, γιατί φαίνεται ότι όσες χώρες είναι κατά, οι χώρες αυτές έχουν τη δυνατότητα πιο εύκολα να τα απαγορεύσουν. Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς απλώς και μόνο απαγορεύοντας την καλλιέργειά τους στην εθνική επικράτεια. Υπάρχει ένας κίνδυνος σήμερα. Και ο κίνδυνος είναι ότι απαγορεύοντας δεν καταφέρνουμε να προστατεύσουμε όπως θα θέλαμε τους πολίτες μας. Γιατί οι γενικά επομένοι οργανισμοί δεν σταματάνε στα σύνορα, ακόμα δηλαδή και αν μια χώρα τους απαγορεύσει, αν μια γειτονική χώρα τους καλλιεργεί, θα φτάσουν και στη δικιά σας. Συνεπώς, το να... Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγουμε την επιμόλυνση αυτή. Θα κοστίζει πάρα πολύ. Εάν λοιπόν η εκμετάλλευση γενετικά τροπημένων οργανισμών γίνει επιτραπή σε κάποιες χώρες, η συνέπεια θα είναι ότι οι οργανισμοί αυτοί θα κυκλοφορήσουν στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης. Άρα τίποτα δεν θα απαγορεύσει την πώληση προϊόντων που περιέχουν τέτοιου γενετικά τροπημένους οργανισμού. Γιατί υπενθυμίζω ότι εδώ η απαγόρευση έχει να κάνει με την καλλιέργεια των οργανισμών αυτών. Άπαξ και οι οργανισμοί αυτοί καταλήξουν σε ένα προϊόν, το προϊόν αυτό θα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. Οι χώρες λοιπόν που δεν θέλουν τους γενετικά τροπημένους οργανισμούς δεν θα, μπορέσουν, δεν θα μπορέσουν να προστατεύσουν τους πολίτες τους όπως θα θέλανε από αυτούς. Και δεν είμαστε καν σίγουροι ότι στις ετικέτες θα υπάρχει υποχρέωση να αναφέρεται το ότι περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Άρα λοιπόν η προστασία των καταναλωτών αποτελεί μια ψευδέστηση, γιατί μία, ένας πολίτης ο οποίος κατοικεί σε χώρα η οποία απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών θα εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνό τους. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι εφόσον την απόφαση την έχουν τα κράτη-μέλη, αυτό θα προχωρήσει κάπως την υπόθεσή μας, θα προστατεύσει περισσότερο τους πολίτες. Δεν λαμβάνουμε δηλαδή με την πρόταση αυτή επαρκώς υπόψη τον κίνδυνο εκείνο ο οποίος οδηγεί τα κράτη-μέλη να μην θέλουν τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Η δυνατότητα λοιπόν που δίνεται στα κράτη-μέλη για απαγόρευση καλλιέργειας γενετικά τροπημένων οργανισμών δεν φτάνει. Δεν είναι αποτελεσματική για την προστασία των καταναλωτών. Εκτός αν προσπαθούσαμε να ενισχύσουμε και τους ελέγχους αν το έργο δηλαδή της ΕΦΣΑ, της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων, γινόταν διαφορετικά. Αλλιώς η Ουγγαρία, η χώρα μου, θα συνεχίσει να πολεμάει τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Και τι θα γίνει, θα απαγορεύσουμε την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην Ουγγαρία, αλλά οι Ούγγροι θα απορροφούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στο σώμα τους, εφόσον η κυκλοφορία τους των οργανισμών αυτών στο εμπόριο θα επιτρέπεται. Ακόμα δηλαδή και αν δεν απαγορευόταν ε, η καλλιέργεια, θα καταλήγαμε λίγο πολύ στο ίδιο. Άρα πρέπει και επιστημονικά και για το περιβάλλον να αξιολογήσουμε καλύτερα τους κινδύνους. Σας ευχαριστούμε Αντιπρόεδρε Γιάβορ και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Πέτυρ για την παρέμβασή του. Της. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήμουν υπέρ του να προταθεί απαγόρευση για τους ε, μη, μη γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς γιατί έχει πλέον αποδειχτεί ότι επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα. Αυτό θέτει λοιπόν σε κίνδυνο ολόκληρο το οικοσύστημα και την παραγωγή τροφίμων. Εάν ε, τελικά εισαχθούν οι οι γενετικοί, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, τότε προσπαθούμε να παραστήσουμε το Θεό είναι κάτι το ανήθικο. Εταιρείε εισάγουν γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και είμαι ευτυχή που η Κροατία είναι χώρα άνευ γάμα όμικρον, γιατί, ε, γιατί κανένας δεν θα πρέπει να μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την απόφαση. δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί αυτού του είδους την βιολογική ε, κυριαρχία της Κροατίας. Πώς μπορούμε εμείς να προστατευτούμε ως χώρα εάν οι γείτονές μας αποφασίσουν να εισάγουν ε, τέτοιους, ε, τέτοιες καλλιέργειες. Αυτό δεν ορίζεται από αυτήν την πρόταση. Ποιος μπορεί να πει, ας πούμε, στις μέλισσες να μην μεταφέρουν γύρι από, δική μας, από μάλλον την άλλη επικράτηση δική μας και αν ε, οι δικές μας καλλιέργειες τελικά επιμολυνθούν, ποιος θα πληρώσει τη νύφη. Τέτοιου είδους ζημιά δεν μπορεί να πληρωθεί με χρήματα. Η Ευρώπη, όπως και άλλες ήπειροι, μπορεί να διατηρήσει την κατάστασή της ως ισορροπημένη ήπειρος από πλευράς ε, περιβάλλοντος και αυτό το θέμα είναι δικό μας, δική μας υπόθεση και ως εκπρόσωπος της Κροτίας θα ήθελα να πω τα εξής. Εάν δεν τροποποιηθεί αυτή η πρόταση θα καλέσω τους γείτονές μας, Σλοβενία, Αυστρία και Ουγγαρία, να, στηρίξει τη δική μου πρωτοβουλία, να στηρίξουν μάλλον τη δική μου πρωτοβουλία που θα ξεκινήσω, ώστε να ε, ε επιβάλλουμε μια ζώνη άνευ γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και να απογορεύσουμε την χρήση αυτών ε, στις επικράτειές μας, προστατεύοντας την βιοπτά μας και το περιβάλλον μας. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Μισελ Ριβαζή για τη δική της παρέμβαση. Εγώ χαίρομαι, Πρόεδρε, που η Ιταλική Προεδρία λέει πως είναι προτεραιότητά της αυτό το θέμα. Αλλά ταυτόχρονα ε, λέω, μα πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Έχουμε καταναλωτές, όπως υπόθηκε, που βασικά είναι κατά της κατανάλωσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Με αυτή τη διαδικασία και θα δούμε πως είναι και τελείως αντιδημοκρατική, προστατεύσαμε την Ευρώπη από την εισβολή των γάμματα φόμικρον. Αν δούμε όμως αλλού τι συμβαίνει, βλέπουμε την κατάσταση της Αργεντινής που είναι καταστροφική με τη χρήση των τα φόμικρον και στην ΕΠΑ δεν υπάρχει ε, γυρισμός και υπάρχει ασυμβατότητα με όσους θέλουν να κάνουν βιολογικά, βιολογικές καλλιέργειες. Εγώ ταυτόχρονα όμως λέω στην Προεδρία πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Έχουμε τον Επίτροπο Γιούνκερ που λέει, έκανε δήλωση και είπε ότι η διαδικασία αποδοχής και αξιοδότησης των γενετικά τροπομένων οργανισμών είναι αντιδημοκρατική. Άρα λοιπόν ας ξαναδούμε την διαδικασία έγκρισης των γάμματα Ε, Έχουμε ειδική πλειοψηφία των κρατών και δεν τα καταφέρουμε. Η Κομισιόν αποφασίζει έναντι των κρατών που είναι κατά των ε, γάμματα φόμικρον. Αυτό είναι δημοκρατικό. Ξαναδείτε αυτήν την ε, διαδικασία και εδώ συμφωνεί και ο Επίτροπος Γιώκερ. Δεύτερον, μιλάμε για αξιολόγηση υγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Η ΕΒΣΑ, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός μας, ε, που επανειλημμένως επικρίθηκε διότι υπήρχαν ε, συγκρούσεις συμφερόντων στο πλαίσιο της ομάδας της. Και όταν έγιναν μελέτες, ο Ντερίκ Σεραλίνη έδειξε ότι υπάρχουν ε, κίνδυνοι ε, υγειονομικοί για ζώα που είχαν καταναλώσει γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο. Είναι αυτό αποδεδειγμένο και η ΕΦΣΑ είχε ε, δείξει ότι, αποδείξει ότι, είχε γίνει αυτή η, ότι υπάρχει μάλλον αυτή η μελέτη. Δεν έχουμε βεβαιότητα και η Μοσάντο κάνει μελέτες, αλλά δεν έχουμε βεβαιότητα όσον αφορά τους, την αξιολόγηση των κινδύνων σε αρουραίους. Κοιτάξτε τι γίνεται στον κόσμο που χρησιμοποιεί αυτούς τους οργανισμούς. Βλέπουμε ότι σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση των σπόρων βλέπουμε κατάρρευση των χωρικών που χρεώνονται μέχρι το λαιμό και από οικονομικής άποψης δεν φέρνει κάτι παραπάνω από ό,τι στις χώρες που δεν χρησιμοποιούν τους γάμματα φόμικρον. Κάντε μια τέτοια μελέτη λοιπόν και βρίσκω ότι ε, αυτή η έκθεση η του Συμβουλίου που εδώ συμφωνώ με τους συναδέλφους και λέω ότι, ότι Τώρα η Κομισιόν, αν ένα κράτος ε, μάλλον αρνείται, θα πρέπει να πάει στην Κομισιόν που θα διαπραγματευτεί με τις εταιρείες, ενώ παλιότερα ήταν άμεσα το κράτος απέναντι στις εταιρείες. Αν μια, ένα κράτος πει όχι, αυτό που δίνετε εσείς ε, είναι νομικός ατελές, γιατί θα μας επιτεθεί ο ΠΟΕ και έπειτα κανείς δεν μίλησε για την ε, Διατλαντική Συμφωνία γιατί αν την υπογράψουμε με τη ΣΥΠΑ και αν υπάρξει αυτό το διαιτητικό δικαστήριο και ότι η χώρα σας, η Κροατία, η Γαλλία, η Αυστρία, οι χώρες μας ε, δεχτούν επίθεση από τη Μονσάντο γιατί δεν μπορούν να έχουν κέρδη και το διοικητικό δικαστήριο μας ζητήσει σημαντικές αποζημιώσεις, τι θα κάνουμε. Θα έχουμε άμεσες επιπτώσεις λοιπόν για την άρνηση ενός κράτους μέλους γιατί θα μπορούν οι εταιρείε να επιτεθούν στο κράτος μέλος. Εγώ είμαι υπέρ μιας ευρωπαϊκής θέσης. Η εθνικοποίηση των κρατών απέναντι στους ε, γάματα, στα γάματα αφόμικρων αν και τη Φρεντερίκ Ρίς την εμπιστεύομαι απόλυτα. Αυτό θα μας τιμωρήσει εμάς τους καταναλωτές και δεν θα έχουμε καμία εγγύηση ότι μέσα στα προϊόντα μας δεν θα έχουμε Γάματα φόμικρον. Προποθέσει, όροι για τη διαδικασία για την αξιολόγηση των κινδύνων για μια κοινωνικο-οικονομική μελέτη, για το, συμφε... το, το, το ενδιαφέρον τη χρήση αυτών των οργανισμών. Α σκεφτούμε του καταναλωτέ, α δούμε τι ε, εκλογέ, εάν δεν σκεφτούμε την προστασία των καταναλωτών και αν δεν ακολουθήσουμε την αρχή τη προφύλαξη, θα χάσουμε πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει ο Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ τις και τους συναδέλφους να είναι μετριοπαθείς στη συζήτηση και να φανούν και ευέλικτοι στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Η κυρία Ζόμερ τόνισε ποια είναι η ισχύουσα νομική κατάσταση. Και, αυτό, και αυτή βρίσκει απήχηση ε, στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Δεν έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα μετά από τις ευρωεκλογέ. Αλλά η κατεύθυνση προς την οποία θα είναι μια δεύτερη ανάγνωση. Έχουμε ισχυρέ δυνάμεις στο Κοινοβούλιο και ιδίως στην πολιτική μας ομάδα που λένε ότι οι αγρότες που θέλουν να καλλιεργήσουν γάμα μειόμικρον ήδη υφίστανται δυσμενή διάκριση λόγω των αποφάσεων του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Παρακαλώ να είμαστε και αντικειμενικοί. Όταν ο αξιότιμος κύριος Γιάβορ των Πράσινων λέει ότι δεν υπάρχει χαρακτηρισμός των γάμα αυτό δεν είναι σοβαρό. Διότι με συμμετοχή και πράσινων υπουργών από διάφορες κυβερνήσεις είχαν εγκριθεί οι σχετικές διατάξεις. Ας μην λέμε τώρα ότι δεν είναι δεδομένη, δεδομένος ο χαρακτηρισμός νομικά δηλαδή. Έχει γίνει αυτό και μάλιστα με μεγάλη ευρύτατη συνένεση. Η κατάσταση τώρα έχει ως εξής. Αν δεν συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, τότε κάθε φύρμα έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει αδειοδότηση, έστω και αν δεν υπάρχει επιστημονική θεμελίωση. Και καθημερινά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενδέχεται να δικαιώνει τις εταιρείες αυτές και το αποτέλεσμα θα είναι να καλλιεργούνται γενετικώ τροποποιημένοι οργανισμοί σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε μέλη. Γνωρίζω ότι είναι, τη δυσκολία της κατάστασης. Όποια και είναι η προσωπική θέση του καθενός για τους γάμματα αφόμικρων, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία σε πολλές χώρες μέλη που δεν τους θέλουν και γι' αυτό εγώ δέχτηκα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι για λόγους οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΕΦΣΑ αλλά άλλους μπορούμε να προχωρήσουμε να δεχθούμε εθνικές απαγορεύσεις. Όμως δεν θέλω να υπάρξει διάσταση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Το Συμβούλιο χρειάστηκε τέσσερα χρόνια και το γνωρίζω αυτό από προσωπικές συζητήσεις με τον Υπουργό μου και με άλλους ότι σε ορισμένε μεγάλε χώρε μέλη, για ορισμένε μεγάλε χώρε μέλη, ήταν πολύ δύσκολο τελικά να δεχτούν το συμβασμό αυτό. Εάν κάνουμε τώρα συζήτηση αρχών και πούμε ότι θέλουμε πανευρωπαϊκή απαγόρευση των γάμματα αφόμικρων, τότε αυτό αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύση. Γι' αυτό και παρακαλώ όλε και όλου του συναδέλφου, ιδίω όμω εκείνου που θα διαπραγματευτούν, κυρία Ρή, είμαι σίγουρο ότι θα δείξετε τον απαραίτητο ρεαλισμό και την απαραίτητη εμπειρία τη διαθέτει τους ή άλλω, ούτε, ούτω ή άλλω και οι σκιώδη συγητές και αυτοί καλούνται να δείξουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε να μην βαθύνει το χάσμα, το οποίο δεν είναι και τόσο δραματικό μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Και να μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λιντίζε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σκόπευα να πάρω το λόγο, λέει η κυρία Γιούσο, γιατί συμφωνώ με την κυρία Σόμερ και τον κύριο Λίσερ, αλλά είναι τόσο σημαντικό θέμα. Μας ε, κάνει όλους να ξεσηκωνόμαστε, έχει να κάνει και με τον επιστημονικό κόσμο και με τον πραγματικό κόσμο, κάτι το οποίο καμιά φορά ξεχνάμε. Υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Πρώτα απ' όλα, η ασφάλεια των γενετικά τροπομένων οργανισμών εξασφαλίζεται. Έχουν γίνει πάρα πολλέ μελέτε. Όταν παίρνει άδεια ένα τέτοιο οργανισμό, σημαίνει ότι είναι ασφαλή. Ό,τι άλλο λέμε δεν ισχύει. Οι προσπάθειε που γίνονται να αποδειχτεί κάτι διαφορετικό δεν είναι αλήθεια και έχει αποδειχτεί αυτό. Έπειτα, η ΕΦΣΑ και οι μελέτες της γίνονται από ανεξάρτητους επιστήμονες. Δεν γίνεται ούτε από την μοντσάντο, ούτε από το διευθυντή της ΕΦΣΑ. Γίνεται από ανεξάρτητους επιστήμονες οι οποίοι έχουν τεράστιο επιστημονικό κύρος, αναγνωρισμένο. Οι ετικέτες. Στο 95% των οργανισμών αυτών υπάρχουν οι ετικέτες, τα προϊόντα δηλαδή που τους περιέχουν εισάγουμε βιομηχανικές ποσότητες τροποποιημένης σόγιας. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να δίνουμε αρκετές πρωτεΐνες στα ζώα μας. Οπότε μπορεί να λέμε ότι θέλουμε για το περιβάλλον κτλ. Αλλά μην λέμε ότι βλάπτουν την υγεία ή ότι θέλουμε να απαγορεύσουμε την κατανάλωσή τους γιατί οι ισοτροφές μας εξαρτώνται από την γενετικά τροποποιημένη σόγια έπειτα για το οικονομικό θέμα όταν καλλιεργούνται είναι γιατί οικονομικά είναι αποδοτικές οι καλλιέργειες αυτές. Ε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, και τώρα ακόμα και αν προχωρήσαμε λίγο περισσότερο από ό,τι είχαμε προβλέψει στη συζήτηση και όλοι θέλαν να εκφράσουν ε, τη θέση τους γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό περνάμε τώρα στην Κομισιόν που πολλές φορές ε, αναφέρθηκε ο κύριος Πουντλέ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πράγματι η συζήτηση αυτή ξεσηκώνει πάντα. Θέλω λίγο σύντομα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόοδο που επετέχθη από την Ελληνική Προεδρία τον Ιούνιο. Η υπόθεση αυτή είχε μείνει πίσω τέσσερα χρόνια. Η πρόταση, μην ξεχνάμε, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2010. Φυσικά και χρειάστηκε να κάνουμε συμβιβασμούς για να μπορέσει το κείμενο αυτό να οριμάσει και να φτάσει στο σημείο που έφτασε στο Συμβούλιο. Θέλω όμως να υπογραμμίσω ότι η πρόταση αυτή για μας προσφέρει μια νομική, επιστημονική ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών. Βελτιώνεται σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. Η σημερινή κατάσταση, όπως γνωρίζετε, μας έχει οδηγήσει σε διάφορες ρήτρε ασφαλείας από τα κράτη-μέλη που νομικά δεν ήταν πολύ και που οδηγούσαν ε, κάποια κράτη-μέλη να καταλήγουν στα δικαστήρια και ο πρόεδρος Μπαρόζο στο πρόγραμμά του, στη δεύτερη θητεία του, θέλησε να εφαρμόσει ένα σύστημα που τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφασίζουν από μόνα τους και να μην είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία να αποφασίζει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επικράτειας όσον αφορά την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η πρόταση αυτή λοιπόν έχει το πλεονέκτημα να προσφέρει νομική ασφάλεια στις χώρες μέλη που θέλουν να μην καλλιεργούν στο εδαφό τους τέτοιους οργανισμούς και είναι οι περισσότερες χώρες, γιατί μόνο πέντε καλλιεργούν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στα εδάφη τους. Η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών δεν θέλει τέτοιες καλλιέργειες. Η νομική ασφάλεια κατά το παρελθόν ήταν ασταθής, αβέβαια και γι' αυτό η πρόταση αυτή ενισχύει την νομική αυτή ασφάλεια σε κοινωτικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Τώρα, Εύσα, επιστημονική ασφάλεια. Εδώ άκουσα διάφορες επικρίσεις για την ΕΦΣΑ. Ε, είναι αλήθεια, πάντα μπορεί κανείς να επικρίνει την Εύσα. Όμως η ΕΦΣΑ εδώ και μερικά χρόνια έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να λύσει τα προβλήματα σύγκρουσης συμφερόντων που είχαν τεθεί. Η επιστημονική αξιολόγηση λοιπόν των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι πιο αυστηρή από ολόκληρο τον κόσμο. Στι ΗΠΑ, στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, έξι μήνε με ένα χρόνο παίρνει η αδειοδότηση τέτοιων οργανισμών. Ενώ εδώ στην Ευρώπη μα χρειάζονται 5 με 10 χρόνια. Και έχει να κάνει αυτό με τι επιστημονικέ αξιολογήσει, οι οποίε είναι πάρα πολύ αυστηρέ στην Ευρώπη. Φυσικά μπορούμε πάντα να τις βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Εννοείται, περάσαμε από δοκιμές ε, τοξικότητας μειωμένης σε άλλες που έχουν να κάνουν με 90 μέρες ε, τοξικότητας και συζητάμε και το θέμα των δύο ετών. Δηλαδή πάντα μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Η κατάσταση όμως σήμερα είναι τέτοια που επιστημονικά είναι η καλύτερη σε ολόκληρο τον κόσμο. Προστασία των καταναλωτών τώρα. Η ΕΦΣΑ μας λέει ότι με τις σημερινές μεθόδους δεν υπάρχει κίνδυνος για τον καταναλωτή. Αν υπήρχε ένας κίνδυνος, τότε θα ήταν τα πράγματα αλλιώς. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν επίσης και συστήματα ε, ετικετών που προβλέπουν στην αγορά ουσιαστικά να μην απολούνται γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, η ανθρώπινη κατανάλωση. Χρησιμοποιούνται μαζικά στις ζωοτροφές. Αλλά όσον αφορά την ανθρώπινη κατανάλωση, πρώτον δεν υπάρχει κίνδυνος και δεύτερον υπάρχει η δυνατότητα ο καταναλωτής να επιλέξει. Αν υπάρχουν ε, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί σε προϊόντα να μην τα αγοράσει. Ακριβώς επειδή αναφέρεται αυτό στις ετικέτες ως επιτοπλίστων. Και υπάρχουν πολύ αυστηροί έλεγχοι στις χώρες μέλη αλλά και στα σύνορα. Αν θέλετε να σας πούμε πώς γίνονται οι έλεγχοι γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, ευχαρίστως να το κάνουμε. Εδώ θέλω να πω και κάτι για το πρώτο στάδιο, το οποίο δεν ήταν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε και σε εκείνη του Κοινοβουλίου, στην πρώτη ανάγνωστη. Προστέθηκε στο Συμβούλιο. Υπήρχαν δύο παράλληλα στάδια και μετά έγιναν διαδοχικά τα δύο στάδια αυτά. Υπάρχει το πρώτο στάδιο και αν δεν λειτουργήσει τότε περνάμε στο δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο έχει το πλεονέκτημα ότι προσπαθεί να διευκρινίσει μια κατάσταση μεταξύ δύο πλευρών και αυτό με, πώς να το με καλό τρόπο, καθώς πρέπει. Μετά οι υπηρεσίες της Επιτροπής σε διαδικασία που βέβαια είναι καθοριστή, Πάντως προς το παρόν η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει ρόλο διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε μια χώρα που αρνείται και μια επιχείρηση η οποία θέλει να καλλιεργήσει τέτοιους οργανισμούς. Προς το παρόν η εκτίμησή μας είναι ότι η Επιτροπή είναι ενδιάμεσος, είναι ένας παράγοντας για να μεταφέρει τη θέση μιας χώρας η οποία δεν θέλει να διαπραγματευτεί με μια επιχείρηση και να τη μεταφέρει στην επιχείρηση αυτή. Όλοι βέβαια ελπίζουν και κυρίως οι επιχειρήσεις γιατί ούτε και αυτές θέλουν ε, ε, διαμάχες. Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα δεχτούν από ό,τι φαίνεται το πρώτο αυτό στάδιο. Εάν δεν λειτουργήσει τότε περνάμε στο δεύτερο στάδιο με την αιτιολόγηση που απαιτείται για να απορριφθεί και νομικά η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ρωτήσατε κάτι για τους διάφορους περιβαλλοντικούς στόχους. Είναι αλήθεια ότι για μας, αν υπάρχουν ε, νέα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά το περιβάλλον, κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, κίνδυνοι για τους ανθρώπους ή για τα ζώα, για τα έντομα, μέλισσες κλπ. Τα νέα αυτά δεδομένα πρέπει να πάνε στην ΕΦΣΑ. Πιστεύουμε ότι δεν είναι καλό μια χώρα μέλη να παίρνει περιβαλλοντικά μέτρα βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα που διαθέτει χωρίς να εμπλέκεται η εύσα. Άλλα περιβαλλοντικά όμως ζητήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αιτιολόγηση όπως είναι η διατήρηση κάποιων φυσικών στοιχείων ή τοπίων, οικότοποι, οικοσυστήματα Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μελετηθούν περισσότερο και στην περίπτωση που υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για μας η ΕΦΣΑ είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ερωτάτε τελικά για το κατά πόσο πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξει η γνωμοδότηση προηγούμενη. Κύριε Πρόεδρε, Αυτά είχα να σας πω για αυτή την πρόταση που εμείς φυσικά και θα θέλαμε να εγκριθεί σε δεύτερη ανάγνωση γρήγορα μάλιστα από την Επιτροπή σας και από το Κοινοβούλιο. Και το θέλουμε αυτό για να μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας ένα κείμενο το οποίο να εγκριθεί οριστικά γρήγορα. Και κάτι ακόμα πριν τελειώσω. έχει να κάνει με τις προτάσεις που έγιναν για τη νέα θέση του μελλοντικού πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Γιούνκερ. Η θέση αυτή είναι νέα. Θα πρέπει να μελετηθεί, να διευκρινιστεί, γιατί πρόκειται για νέα στοιχεία που έβαλε στο τραπέζι, προκειμένου να μπορούμε να σεβαστούμε την άρνηση αυτή των πολιτών μας για γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Πρέπει να ξέρουμε ότι η γεωργία εξαρτάται πάρα πολύ σήμερα από την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και ε, πράγματι αν η γεωργία δεν μπορεί να έχει στη διάθεσή τη τέτοιου οργανισμούς για να ταΐζει τους χείρους, τις αγελάδες, τα πουλερικά κτλ, αυτό οικονομικά θα είχε τεράστιο κόστος. Πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο οικονομικό κόστος για να μην έχουμε γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Αυτή είναι τεράστια πολιτική απόφαση, την οποία βέβαια το Κοινοβούλιο θα πάρει ενδεχομένως, ζυγίζοντας τα υπέρ και τα κατά. Πάντως εμείς με τον επόμενο αρμόδιο επίτροπο και τον πρόεδρο Γιούγκερ θα εξετάσουμε την αυτή πολιτική για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πουτλέ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βεντουρέλη, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ όλους για αυτή τη συζήτηση που ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Νομίζω τουλάχιστον εννέα σελίδες ε, σημειώσεις έχω κάνει με συγκεκριμένα και πιο γενικά με τα ερωτήματα και σίγουρα θα προσπαθήσω να απαντήσω ε, σε όσο περισσότερες ερωτήσεις ε, τέθησαν ε, και τις υπόλοιπες μετά από όταν θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Να ήθελα όμως να απαντήσω σίγουρα σε κάποιες ερωτήσεις από τώρα γιατί κάποιοι εξέφρασαν σχεδόν απόγνωση για την ένταξη της πρώτης φάσης στον μηχανισμό opt-out. Η πρώτη φάση όμως δεν θέλει να είναι φάση διαπραγμάτευσης με την εταιρεία. Όπως είδαμε τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε ότι ορισμένε εταιρείε αποσύρουν τα αιτήματα αδειοδότησης. Η πρώτη φάση θέλει να δώσει νομική βεβαιότητα με ξεκάθαρο τρόπο από την αρχή της διαδικασίας. Ένα αίτημα που υποβάλλεται από το κράτο μέλος μέσω της Κομισιόν προς την εταιρεία ε, δεν είναι διαπραγμάτευση. Η εταιρεία μπορεί να πει όχι, οπότε ε, ξεκινάει η δεύτερη φάση ε, και με συγκεκριμένα προθεσμίες, αλλά στην περίπτωση που δεν πει τίποτα, σημαίνει πως εξ αρχής θα υπάρχει νομική βεβαιότητα για όλους τους φορείς, για τα κράτη-μέλη και για τους ε, ε, ε, φορείς, γιατί ο γεγονός ότι η γεωγραφική κάλυψη, το γεωγραφικό εύρος είναι περιορισμένο. Και αυτό έτσι ώστε να πούμε ότι χρειάζεται, και άκουσα μάλλον από εσάς ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία, μα αυτή είναι η ευελιξία που, στην οποία κατέληξαν τα κράτη-μέλη στο, τελευταίο ε, Συμβούλιο. Ε, ακριβώς ε, έτσι ώστε να διευκολύνουν και τα επόμενα βήματα. Είναι αλήθεια πως η συζήτηση και η κοινή γνώμη είναι όλοι πολύ έτσι, τεταμένη η κατάσταση. Όλοι θέλουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα και ο στόχος δεν είναι δυστυχώς ή ευτυχώς να αλλάξει το σύστημα αδειοδότησης, το κοινοτικό σύστημα αδειοδότησης. Όπως γνωρίζετε, αυτό εξαρτάται από το τι θα κάνει ενδεχομένως ο πρόεδρος Γιούνκερ και ε, με την νομοθετική πρωτοβουλία που προέρχεται από την Κομισιόν και γι' αυτό και πρέπει να περιμένουμε πρόταση της Κομισιόν. Αλλά για να λυθούν τα άμεσα προβλήματα που όλα τα κρατημέλη συναντούν, Θεωρούμε ως ε, Προεδρία και ως Συμβούλιο πως είναι σημαντικό να ενεργήσουμε άμεσα και να δώσουμε στα κρατημέλη τη δυνατότητα να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την χρήση. Ε, είναι σημαντικό ότι αυτό το κείμενο το συμβιβαστικό που ορισμένοι το επικρίνατε, άλλοι λιγότερο, ε, εγκρίθηκε από 27 κράτη-μέλη. Ε, ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχουν 20-21 που ε, κατά βάση είναι κατά της καλλιέργειας των ε, γάμα ταφ όμικρον. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ότι θα πρέπει να υπάρχει επαρκής νομική ασφάλεια, νομική βεβαιότητα για να μπορεί κανείς μετά να ενεργήσει σε εθνικό επίπεδο. Ε, βεβαίως η συζήτηση είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσα και θα υπάρχει ε, τρόπος να το συζητήσουμε και αργότερα, να μιλήσουμε για την νομική βάση, για την οικονομική ευθύνη, για συντελεστές, για συνύπαρξη. Ξέρουμε ότι είναι θέματα για τα οποία το Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένες θέσεις. Πάντως όσον αφορά τα, τα αίτια μπορούμε να αποφασίσουμε να το συζητήσουμε. Εγώ δεν έχω τέτοια διαπραγματευτική εντολή και σίγουρα δεν μπορώ να πω κάτι σε σχέση με αυτόν τον κατάλογο, πάντως σίγουρα είναι ένας ανοιχτός κατάλογος, ακριβώς για να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ευελιξία αυτός ε, θεωρούμε ότι είναι και ο στόχος αυτής της πράξης, δηλαδή η ευελιξία και η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν καταστάσεις όπως αυτή που τώρα δημιουργεί προβλήματα. Ελπίζω πως αυτός θα είναι και ο στόχος του Κοινοβουλίου και είμαι βεβαία ότι θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε με αποτελεσματικό τρόπο με την κυρία Ρή, και όλους οδησυσυγητές και όλους σας, ώστε να φτάσουμε σε συμφωνία μέχρι το τέλος του χρόνου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ε, κυρία Βεντουρέλη και συνήθως τη συζήτηση κλείνει η συγγήτρια με μια παρέμβασή της. Δεν ξέρω αν θέλει να απαντήσει η συγγήτρια ή να προσθέσει κάτι ή αν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί ε, έχουμε τελειώσει και το χρόνο μας. Να προσθέσω μόνο ότι με τη διαβίβαση της ε, κοινής θέσης του Συμβουλίου στην ε, Σύνοδο του Σεπτεμβρίου το επόμενο, η επόμενη προθεσμία θα είναι η εξέταση τη σύσταση στην ΕΜΒΗ από τον 9 Οκτωβρίου, προθεσμία για τις τροπολογίες 14 Οκτωβρίου και διαπραγματευτική εντολή στις 5 και 6 Νοεμβρίου και στη συνέχεια η ψηφοφορία πρώτα στην Ολομέλεια της ΕΜΒΗ και μετά στην Ολομέλεια τον Γενάρη. Τώρα όμως έχουμε αργήσει πολύ να πω σε σχέση με το ωράριό μας. Είχαμε ζητήσει από τον συνάδελφο Γκέρμπερ αν μπορούμε το θέμα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να το εξετάσουμε το απόγευμα αφού θα έχουμε ακούσει τους δύο επιτρόπους αλλά έχουμε Του εκπροσώπου τη Κομισιόν που ήρθαν από το Λουξεμβούργο για να μα ενημερώσουν για την κατάσταση εργασιών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το αλκοόλ. Και να δούμε πώ μπορούμε γρήγορα να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Και να δώσω αμέσω λοιπόν το λόγο στον συνάδελφο Βίλμοτ, στην συνάδελφο Βίλμοτ που πρότεινε αυτή την πρωτοβουλία και μετά στην Κομισιόν για να κάνει την παρέμβασή της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το θέμα σημαντικό και καλό θα ήταν να τηρούν σιγή ε, αποχωρούσε και οι αποχωρούντες. Και είναι κρίμα που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε. Παρακαλώ ησυχία. Για να μπορέσετε να ακούσετε τη συνάδελφο και μετά την Επιτροπή. Όσοι θέλετε να φύγετε από την αίθουσα να φύγετε, αλλά παρακαλώ ευγενικά και σιωπηρά. Ευχαριστώ. Όπως είπα είναι σημαντικό το θέμα. Όλοι και όλες αντιλαμβανόμεθα ότι οι σοβαρές επιπτώσεις μάλλον τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει το ενόπνευμα στην υγεία. Και έχουμε και πολλές επιτυχίες από την πολιτική για το ενόπνευμα. Παρακαλώ κάντε κάποια ησυχία. Παρακαλώ να καθίσετε. Προέδρο, σου παρακαλώ το Συμβούλιο, αν ε, έχετε να μιλήσετε, να πείτε κάτι, κάντε το έξω παρακαλώ. Ε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, δεν μας έχει δοθεί πρόταση για νέα στρατηγική για το αλκοόλ. Κανένας δεν έχει δει πρόταση ακόμα. Δεν έχουμε καμιά διαβεβαίωση ότι θα ανανεωθεί παρά σαφή πίεση από το Κοινοβούλιο και τα κρατημέλη. Αν ανανεωθεί μάλλον θα είναι για το 2016 με 2022 και... Ε, τελευταία σχετικά σχετική απόφαση ε, διερκούσε μέχρι το 2012. Ε, εγώ θα θέλω να εξασφαλίσω ότι θα αρχίσουμε να εργαζόμαστε για αυτό το ψήφισμα όσο γίνεται ε, πιο γρήγορα, μάλιστα άμεσα και θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στο Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Και για το δεύτερο θέμα, την έκθεση για την τικετοθεσία για το αλκοόλ θα έπρεπε να έχει γίνει και δεν έχουμε δει κάτι σχετικό. Αντίθετα με άλλα προγράμματα τα, οι ετικέτες των ε, υπνοπνευματοδών δεν συμπεριλαμβάνουν καμία πληροφορία όσον αφορά τις βασικές πληροφορίες για τη διατροφή. Το ίδιο είπαμε για τη σοκολάτα και η παχυσαρκία και άλλα σχετικά προβλήματα που είναι πολύ σημαντικά και θέλουμε ε, να ξέρουμε πότε θα έχουμε και αυτή την έκθεση. Παρακαλώ, θέλω απαντήσει. Σα ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα δύο που ζήτησαν το λόγο και παρακαλώ το συναδέλφου να είναι σύντομοι και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Ντάνκαν. Ευχαριστώ. Έχω κάποια θέματα. Η ίδια η προηγούμενη στρατηγική για το ενόπνευμα είχε κάποιες, έδειξε κάποιες επιτυχίες. Να μην χάσουμε λοιπόν τις πρόοδους που επιτεύχθηκαν μέσω κίνηση της στρατηγικής. Το ίδιο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το one size fits all δεν μπορεί να είναι σωστή απάντηση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές και εθνικές διαφορές στα θέματα που έχουν σχέση με το ενάπνευμα. Συμφωνώ με τα σχόλια για την επισήμανση των ε, ενόπνευματοδών. Πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς τι καταναλώνουν. Καθώς βεβαίως και το περιεχόμενο σε θερμίδες. Η πρόκληση για τη νέα στρατηγική θα είναι να συμμορφώνεται με τις βέλτιστες πρακτικές, με τις συνήθειες των χωρών μελών και να αποδίδει. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό, αλλά μέχρι τώρα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και δεν εξυπηρετεί την αξιοπιστία των άλλων θεσμικών οργάνων. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει κάποια πρόοδο και μάλιστα σύντομα για να διασφαλίσουμε ότι το σημαντικό αυτό θέμα θα ξαναλάβει κάποια κίνηση. Μάλιστα κύριε Σουίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη την προηγούμενη φορά είχα ζητήσει το λόγο για την στρατηγική για το ενόπνευμα βρίσκω ότι είναι κρίμα που ακόμη δεν έχουμε αρχίσει να επεξεργαζόμαστε τη νέα στρατηγική για το ενόπνευμα. Έχει λήξει τώρα πλέον το στρατηγικό σχέδιο του 2012 και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει να επεξεργόμαστε το νέο. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε. Διότι υπάρχουν όντω πολιτιστικέ διαφορέ, τι οποίε πρέπει κανεί να λάβει υπόψη, αλλά αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Η επισήμανση είναι σημαντική, η ένδειξη για τις θερμίδες είναι σημαντική και είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι ένα ποτήρι κρασί έχει τον ίδιο αριθμό ε, θερμίδων όπως μια πλάκα σοκολάτα. Βεβαίως υπάρχουν και οι διαφορές μεταξύ βορρά-νότου. Οι παραδόσεις είναι διαφορετικές. Σε ορισμένες χώρες μέλη μάλιστα το ενόπλα θεωρείται και τρόφιμο. Απ' την άλλη μεριά για τους νέους συχνά αποτελεί πάθος. Χρειάζεται λοιπόν να αναπτυχθεί μια στρατηγική η οποία να τηρεί και τους θεμελιωδέστερους κανόνες. Σας ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν ώστε να μπορέσει να μας ενημερώσει για το ποιε είναι οι διαθέσεις της όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το αλκοόλ. Um, ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο παρά το προχωρημένο της ώρας. Θέλω να αντιδράσω λίγο αναφέροντας πρώτα απ' όλα, έχοντα ακούσει και τα σχόλια των Ευρωβουλευτών, ότι η αντίληψη που έχετε ότι δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι το 2012, ίσως να είναι κάπως λάθος. Γιατί? Γιατί έχουμε αξιολόγηση της στρατηγικής με εξωτερική αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε το 2013 και κατέληξε σε ένα ενδιαφέρον συμπέρασμα το οποίο ήταν ότι τα μέσα, τα εργαλεία που διαθέτει από το 2006 η, η προσπάθεια αυτή είναι ικανοποιητικά. Οπότε το ερώτημα τίθεται τότε τι εφόσον το μόνο ζήτημα που υπήρχε και υπάρχει ακόμα είναι ότι παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα εξακολουθούμε να έχουμε υψηλά επίπεδα κατάχρησης. Προσπαθούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα να επενδύσουμε περισσότερο στα μέσα τα οποία έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Και συμφωνήσαμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στόχος του 2006 εξακολουθεί να ισχύει, θα έπρεπε να συνεργαστούμε με τις χώρες μέλη και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για να διασφαλίσουμε και αποτελέσματα. Δουλέψαμε λοιπόν με την ε, Επιτροπή όπου συγκεντρώνονται οι εθνικοί φορείς για να δούμε με ποιο τρόπο θα πετύχουμε πιο γρήγορα. Μαζί τους λοιπόν και με τις χώρες μέλη δουλεύουμε εδώ και μήνες για να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα δράσης των κρατών μελών όσον αφορά την ε, κατανάλωση αλκοόλ. Εδώ είναι που τα κράτη-μέλη θέλουν γρήγορα κάποια πρόοδο. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα, δώσαμε και οικονομική στήριξη για κοινέ δράσεις των κρατών μελών, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα όπου τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους και να έχουν παρετέρω δράσεις. Και καταλήξαμε ότι και αυτή η κοινή δράση και το πρόγραμμα δράσης αποτελούν σημαντικά εργαλεία για να καταλήξουμε στο κατά πόσο χρειάζεται μια νέα στρατηγική ή η στρατηγική του 2006 φτάνει. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπούμε σε ένα πλαίσιο δράσης. Σήμερα λοιπόν δεν είμαι σε θέση να σας πω κατά πόσο θα υιοθετήσουμε νέα στρατηγική ή όχι. Αυτό που είναι όμως σαφές είναι ότι θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη ώστε να δούμε ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος να προχωρήσουμε. Στρατηγική. Ίσως και κάτι άλλο που ίσως σας ενδιαφέρει είναι ότι διευκολύνουμε στην ΑΠΑ το έργο των χωρών μελών Και αυτό ακριβώς θα αποτελέσει και τη βάση για συζήτηση με την Επιτροπή για το ποιο θα μπορούσε να είναι το μέλλον μιας νέας στρατηγικής. Γιατί μια νέα στρατηγική σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και κάτι καινούριο, κάτι άλλο. Αν συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα, τότε θα ε, επρόκειτο απλώς και μόνο για μια ανανέωση του υπάρχοντος πλαισίου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μακρηγορώ. Αν θέλετε κάποια άλλη στιγμή να σας δώσω περισσότερα λεπτομέρειες για το σχέδιο δράσης όταν θα έχει εγκριθεί από τα κράτη-μέλη και αφού έχουν συζητήσει τα κράτη-μέλη μεταξύ τους περισσότερο. Ευχαριστώ. Wilmot. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν αρκούν αυτά. Είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο θέλει στρατηγική για το μέλλον και δεν είναι αρκεί να μας λέτε το κάναμε, το είδαμε το περασμένο χρόνο και δεν έχουμε κάνει τίποτα έκτοτε. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να δούμε τις minimum ε, τιμές, θα μπορούσαμε να δούμε ε, τις περιορισμούς ε, στη διαφήμιση κτλ. Ένα σωρό πράγματα να αυξήσουμε επίσης ε, τα χρήματα για την έρευνα. Ε, ε, θέλουμε πάντως κάτι να γίνει και να αντικαταστήσει τη στρατηγική. Διαφορετικά θα χάσουμε την κατάλληλη στιγμή. Πρέπει να επανέλθετε με κάτι κάπως πιο συγκεκριμένο και μην μας λέτε μόνο μην ανησυχείτε το εξετάζουμε. Δεν μας αρκεί αυτό. Πρόεδρος, εγώ Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω την Κομισιόν για αυτή την παρουσίαση. Σίγουρα μετά το Κοινοβούλιο σε επόμενες διαδοχικές ευκαιρίες θα λάβει τις αποφάσεις του και θα ορίσει τη θέση του. Για το θέμα, σε μια από τις επόμενες μας συνεδριάσεις. Ευχαριστώ την Κομισιόν και θα τα πούμε αργότερα για να συνεχίσουμε τις απογευματινές εργασίες.